Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλες. Φίλες και φίλοι μάλλον. Φίλες και φίλε, λέει ο πρόεδρος. Επαναλαμβάνεται η σύνοδος. Έχουμε μεταξύ μας την Επίτροπο και συνάδελφο Μάλστρεμ και θα ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα της μύρισιας διάταξης που είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Ζαν Λαμπέρ για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, θέμα ύψης της σημασίας. Γιατί η κυρία Λαμπέρ θα μας ε, διευκρινίσει την κατάσταση μας, την εκθέση μάλλον. Κυρία Λάμπερτ, έχετε τέσσερα λεπτά για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ε, εμπνεύσω. Πρόκειται για θέμα για το οποίο υπάρχουν πολλές διαφωνίες, ε, για το οποίο πολλά μέλη του Κοινοβουλίου θα φοβούνταν να μιλήσουν γι' αυτό. Οπότε οι γενναίοι που βρισκόμαστε εδώ πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ ενεργό συμμετοχή τους και την δυνατότητα που μας έδωσαν να βρούμε μια κοινή διαπραγματευτική θέση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο προεδρίες, Τσεχική και Σουηδική, για την πιο ανοιχτή προσέγγιση που είχαν σε σχέση με παλαιότερες διαπραγματεύσεις, όπου όντως μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε σχετικά ελεύθερα και όχι απλά να αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό που ήθελε το Συμβούλιο, τουλάχιστον όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Ο στόχος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι να έχουμε μια συνεκτική διαδικασία για αυτούς που χρειάζονται προστασία και πρόκειται για θέμα ζωής και θανάτους για όσους ε, έχουν ανάγκη από αυτή την στήριξη. Όμως υπάρχουν πολλές διαφορετικές μεταξύ των κρατών μελών μεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για όσους προσπαθούν να λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις και βεβαίως τελικά κάποιοι εξαιτία εξαιτίας αυτού. Επίσης ορισμένα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό δυσανάλογη πίεση αισθάνονται ότι δεν υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη και ότι δεν χρειάζεται κάποια πρακτική απάντηση. Στα πλαίσια του Ταμείου Προσφύγων έχει υπάρξει κάποια συνεργασία συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που έχει οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις. Έδειξε όμως ότι υπάρχουν και περιορισμοί σε αυτή την προσέγγιση. Οπότε υπάρχει δέσμευση πλέον να έχουμε μία ενεργή στήριξη για τις χώρες που βρίσκονται υπό δυσανάλογη πίεση και για μεγαλύτερη συνεργασία. Τα βασικά στοιχεία για το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις ήταν καταρχάς ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την υπηρεσία υποστήριξη για το άσυλο, η μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, καθώς και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και του UNHCR. Αυτά τα είδαμε σε σχέση και με την διορισμό του Διευθυντή και του Συμβουλίου και της Επιτροπής υπήρξε μία εμπιστευτική γνωμοδότηση και προσπαθήσαμε να λάβουμε πληροφορίες σε σχέση με αυτό. Επίσης, χρειάστηκε να πιέσουμε για να έχουμε ετήσια έκθεση και θα μπορεί ο διευθυντής να προσκαλείται στο κοινοβούλιο για να μας ενημερώσει για συγκεκριμένα εργασίες της υπηρεσίας υπάρχει μια διοργανική ομάδα εργασίας που ασχολείται με το θέμα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής εκ μέρους του Κοινοβουλίου που διαπραγματεύεται το θέμα. Περνάω στην αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο ήθελε δεσμευτικά μέτρα, το Συμβούλιο ήθελε εθελοντική συνεργασία, τελικά η διατύπωση είναι περισσότερο ουδέτερη. Πάντως, το θετικό είναι ότι θα έχουμε εξωτερική αξιολόγηση που θα εξετάζει την, τον αντίκτυπο της υπηρεσίας στην πρακτική συνεργασία για το άσυλο. Όσον αφορά το φόρουμ, για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Προφανώς υπάρχει μεγάλη εμπεριγνωμοσύνη στα κράτη-μέλη που θα μπορούσε να ήταν πολύτιμη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν σχέσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μας ενδιαφέρει αυτό και επίσης μας ενδιαφέρει και η σχέση με τις τοπικές αρχές οι οποίες θα είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή του συστήματος. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτές να συμπεριληφθούν. Χαιρόμαστε που έγινε κάτι τέτοιο και έτσι ζωντάνεψε περισσότερο η υπηρεσία. Τελικά, θεωρούμε ότι μπορούμε να παίξει σημαντικό ρόλο η υπηρεσία για το άσυλο στην δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο και στην ε, ενίσχυση της συνεργασίας και της δημιουργίας μια κοινή ατζέντα για το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ζητήσω από τα κράτη-μέλη να είναι πιο ανοιχτοί και να συμμετέχουν περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπορούν να συμμετέχουν άλλοι φορείς και η κοινωνία των πολιτών. Γιατί αυτό το θέμα δεν είναι μόνο διακυβερνητικό. Έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα νέο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Η κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση την ανακοίνωση και εισήγηση της, συντάκτρια, της συντάκτριας χαίρομαι διότι θα εγκρίνουμε τελικά τον κανονισμό για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας ασύλου. Είχε προταθεί το Φεβρουάριο του 2009 και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δεσμευτεί επ' αυτής. Η θέσπιση ενός κοινού συστήματος ασύλου ήταν στόχος εδώ και πολλά χρόνια και η Επιτροπή καθώς και εγώ έχουμε δεσμευτεί προς αυτό. Θα πρέπει να προωθήσουμε ένα δίκαιο σύστημα με βάση κοινέ αρχές και να βασίζεται βεβαίως και στην αλληλεγγύη με τους μετανάστες, με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης, ε, αλλά και με όλα τα κράτη-μέλη. Για να ενισχύσουμε την ε, αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών χρειάζεται έμπρακτα συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών για να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό σύστημα ασύλου και για να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία χρειάζεται ένα γραφείο υποστήριξης όπως ζητήθηκε το 2008 με βάση την ε, πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και εγκρίθηκε από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης του 2009. Αυτό είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινή πολιτικής ασύλου. Όπως ξέρετε θα συσταθεί, ε, θα έχει έδρα την ε, Λαβαλέτα και θα προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μέσα στα πλαίσια κοινών πρακτικών με κοινέ πρακτικές, έγκριση και έλεγχο ετοιμάτων χορήγησης ασύλου και ούτω καθεξής. Επίσης, το Γραφείο Υποστήριξης θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη με ομάδες εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με τα αιτήματα των κρατών μελών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους συζητητές που ήταν υπεύθυνοι και βεβαίως την κυρία Τζιν Λάμπερτ για την εξαιρετική της εργασία και τον κύριο Μόρες για τις τροπολογίες καθώς και τους σκιώδεις και κοινούς συντάκτες. Η συνεχή σας υποστήριξη ήταν, είναι μνημόνευτη και ελπίζω ε, πολύ σύντομα να συσταθεί αυτό το γραφείο ε, υποστήριξη. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Μπαίνουμε στους, ε, στους ομάδες ομιλητών, στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Ο κύριος Μπουζούτιλ έχει το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Λάμπερτ για την έκθεσή της και για την επιτυχία που σημείωσε ως προς αυτό το θέμα. Συνεργάστηκε με όλους τους κοιόδης και το ΕΛΚ θα τηρήσει πολύ θετική στάση ως προς την ίδρυση αυτής της υπηρεσίας γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό βήμα τη δημιουργία της υπηρεσίας για την καλύτερη στήριξη των αιτητών ασύλου και τη προς πρώτο βήμα μιας κοινή πολιτικής ασύλου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, είμαι περήφανος ως Μαλτέζος βουλευτής ότι στη, διότι στη Βαλέτα θα εδρεύει η υπηρεσία αυτή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου πρέπει να βασίζεται σε μία και μόνο λέξη αλληλεγγύη η οποία πρέπει να επιδεικνύεται προς εκείνους που έρχονται στην Ευρώπη ζητώντας άσυλο και που έχουν δικαίωμα να δεχτούν κάποια, να πάρουν κάποια προστασία από την Ευρώπη. Αυτό θα διασφαλίζει η υπηρεσία αυτή και επίσης αλληλεγγύη με τις χώρες που όπως είπε και η Επίτροπος, με τις χώρες μέλη στην Ένωση που αντιμετωπίζουν από μόνες τους αυτό το πρόβλημα και το βάρος αυτό δεν μοιράζεται όπως θα έπρεπε. Η αλληλεγγύη λοιπόν αυτή πρέπει να εννοηθεί με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Διπλή αλληλεγγύη με τους αιτητές σύλλου και με τις χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο βάρος και πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το, το μήνυμα αυτό πρέπει να πω ότι έχει γίνει κατανοητό φαίνεται. Αλλά πρέπει τώρα να μεταφραστεί και στην πράξη. Και εδώ βρίσκεται ο ρόλος και η θέση αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου. Εκεί θα φανεί αν η αλληλεγγύη όντως μεταφραστεί στην πράξη, αν, υπάρχει, αν υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη. Ελπίζω λοιπόν η υπηρεσία αυτή να αρχίσει τις εργασίες της όσο το δυνατόν συντομότερα και θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι ως ευρωβουλευτές θα παρακολουθούμε στενά και τους μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν την λειτουργία του. Θα ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε σε οικογενειακή σύνθεση, να τηρείτε το χρόνο σας για να μην σας ε, διακόπτω. Εν πάση περιπτώσει έχετε αρκετό χρόνο ως ομάδες. Από τους σοσιαλιστές η κυρία Σιλβίγη έχει το λόγο για τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Λαμπέρτ και τον κύριο Μωράης για την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσαν και όταν αποκατασταθεί η τάξη στις εναέριες κυκλοφορίες θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα δημιουργίας του Γραφείου Υποστήριξης. Είμαστε ομόφωνοι ως προς τη δημιουργία αυτού του Γραφείου Υποστήριξης. Επειδή θα πρέπει να προωθήσουμε την άμεση συνεργασία θα πρέπει να πληρώσουμε τα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών για τη δημιουργία του ασύλου. Έτσι ώστε να προωθήσουμε την εναρμόνιση που άρχισε με το Τάμπερε. Θα πρέπει να υπάρξει συνοχή και θα ήθελα να τονίσω και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών μέσα στα πλαίσια των συμβουλευτικών φόρουμ. Θα προωθήσουμε με επιτόπιες δράσεις ε, τις διασαφήσεις που χρειάζονται σε θέματα ασύλου και θα καλύψουμε και τα εθνικά ελλείμματα. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα λυπηρά στοιχεία, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να ε, επηρεάσει τον διορισμό του Διευθυντή του Γραφείου. Και επίσης μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης, η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μεταξύ κρατών μελών για να βοηθήσουμε τις χώρες, τις όμορες χώρες δεν μιλάμε για ένα πλέον πιο δεσμευτικό σύστημα, πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Το θέμα είναι επίκαιρο και θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε στους συνομιλητές μας, Επιτροπή και Συμβούλιο. Μιλάμε για ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Μιλάμε για δηλώσεις όπως αυτό της, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου του 2008, όμως ε, ορισμένοι πλήττονται από αμνησία όταν πρόκειται να περάσουμε σε πράξεις και σε κοινού κανόνες. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο με μεγάλη σπουδή έχει εγκρίνει θέματα για την αντιμετώπιση της ε, παράνομης μετανάστευσης, αλλά δεν έχει ασχοληθεί με το πακέτο ασύλου, έτσι ώστε να προωθήσουμε μέτρα τα οποία να μην είναι κατασταλτικά. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη να προωθήσουν μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Τα κατασταλτικά μέτρα δεν βοηθούν στη χορήγηση ασύλου, γιατί γίνονται πολλά ε, κοσκινίσματα και τα ταξίδια γίνονται πιο επικίνδυνα θα πρέπει να μιλήσουμε για εναρμόνιση διαδικασιών χορήγησης ασύλου με πραγματικές εγγυήσει για τους ετούντες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αντίσταση από τα κράτη-μέλη και προωθούν εθνικές, προ... Ε, εθνικές ε, ε, θέσεις και οπτική γωνία. Νομίζω ότι αυτό όμως είναι απαράδεκτο στα πλαίσια και της παγκόσμιας κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι πολλές ε, τρίτες χώρες έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους έναντι της χορήγησης ασύλου. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε και με το γραφείο υποστήριξη. Ευχαριστούμε για δυόμιση λεπτά. Η κυρία Βεριζά από την ΚΟΕ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι από τα βασικά δικαιώματα της Ένωσης και κανείς δεν μπορεί δημόσια να το αφισβητήσει. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη βλέπουμε ότι τίθενται αμφιβολίες από ορισμένα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικά χρόνια άρχισε να εναρμονίζει την πολιτική ασύλου της και κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των αιτητών. Και εμείς στην ΚΟΕ χαιρόμαστε για αυτό, θα χαιρόμασταν εάν αυτό σήμαινε ότι μειώθηκε το πρόβλημα. Όλοι όμως και όλες γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι συζητήσεις μας τις πέμπτης απόγευμα το δείχνουν. Πρόκειται για εναρμόνιση προς τα κάτω των διαδικασιών που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των αιτητών και κάθε χώρα ε, ακολουθεί διαφορετικούς δρόμους Ορισμένοι που ζητούν άσυλο δεν μπορούν, έχουν καν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει δείξει τη χειρότερη συμπεριφορά και επειδή εγώ είμαι αγωνίστρια στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξέρω τι λέω, αρκεί να πάει κανείς έστω και μία φορά να ακολουθήσει τι, τι πρέπει να κάνει ένας αιτητής ασύλου για να δει τι αντιμετωπίζει. Τους ζητούν αποδείξεις για τα βασανιστήρια που έχουν υποστεί και αυτό είναι απαράδεκτο. Η σημερινή μας λοιπόν έκθεση είναι κάτι το πολύ θετικό γιατί συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης και τη προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος για το άσυλο και μιας, ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών με καλύτερη πρόσβαση των πληροφοριών από τις διάφορες χώρες. Και αυτό είναι θετικό. Οι περισσότερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και γνωρίζουμε ότι αυτό το οφείλουμε ιδιαίτερα στην Σουηδική Προεδρία, την οποία και ευχαριστούμε. Προσθέτω ότι η Σουηδία για μένα είναι πρότυπο και υπόδειγμα και θα ήθελα και άλλες χώρες να την ακολουθήσουν. Στην πρώτη ανάγνωση αλλά και στη δεύτερη Υποστηρίξαμε την συγκήτρια και την συγχαίρω και εκείνη, καθώς και την ευχαριστώ. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Ολομέλεια και θα θέλαμε η μικρή αυτή πρόοδος να αποτελέσει καμπή στην ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο αντί να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να δημιουργούμε την λεγόμενη Ευρώπη Φρούριο θα έπρεπε να δεχτούμε στην αγκαλιά μας αυτούς τους ανθρώπους και των δύο φίλων έτσι ώστε να σεβόμαστε και την ε, Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξ ονόματος της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Μποργκέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα το θέμα της αλληλεγγύης. Αυτό επικαλεστήκατε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι και η ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θεωρούμε ε, αυτά τα θέματα. Εγώ έχω ταξιδέψει πολλές φορές με τους ε, καραμπινιέρι και άλλες συνοδευτικές ομάδες του Τωρίνου και μου είπαν ότι πολλές φορές οι ετούντες άσυλο παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία και έγγραφα. Θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή του θέματος, δηλαδή το θέμα της ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι αυτό το έγγραφο καλύπτει την πτυχή της ασφάλειας επαρκώς. Και όμως είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί δεν θα πρέπει να μολύνουμε ε, μία αρχή, μία βασική αρχή δηλαδή της χορήγησης ασύλου με βρώμικα συμφέροντα, δηλαδή αυτών που προωθούν ε, την παράνομη μετανάστευση για καθαρά βρώμικους σκοπούς, δηλαδή για το άνομο κέρδος. Το άρθρο 2 του κανονισμού αναφέρει ότι το γραφείο θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να προωθήσουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου, ακόμα και όσον αφορά την εξωτερική ε, πλευρά. Και το άρθρο 5 αναφέρεται σε αυτό, αλλά χωρίς αφήνεια. Δηλαδή μπορεί να προωθήσει μορφές συνεργασίες ε, με τρίτες χώρες για τεχνικά θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα. Γιατί δεν προτάθηκε η σύσταση αυτών γραφείων υποστήριξης και σε τρίτες χώρες. Τι δεν, γιατί δεν μας επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελαφρύνουμε τον φόρτο εργασίας και θα πρέπει να υπάρχει μια μεσότητα από τις τρίτες χώρες, διότι θα πρέπει να ναι. τύχουν υποστήριξη σε αυτές οι χώρες. Νομίζω ότι χρειάζεται η σύσταση ε, γραφείων και σε τρίτες χώρες, δηλαδή στην υποσαχάρια περιοχή, στη Βόρεια Αφρική, από όπου προέρχονται πολλά αιτήματα. Θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και η υπηρεσία μας εξωτερικών σχέσεων και διπλωματικών σχέσεων με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να τους θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους. Νομίζω ότι αυτές οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές και δεν πρέπει να τις απαρνούμεθα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις απαιτήσει των κρατών μελών της Μεσογείου. Έχουμε πολλούς γραφειοκράτες ήδη. Χρειαζόμαστε χρήματα, χρειαζόμαστε κονδύλια, μέσα, πραγματικά μέσα υποστήριξη. Γιατί εντάξει, στη Σουηδία έχουν ε, καλό στα πράγματα, αλλά είναι διαφορετικά η κατάσταση στη Μεσόγειο, στη Μάλτα, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εφόσον έχουμε εμείς την ευθύνη θα πρέπει να βρούμε και τα μέσα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μποργέζιο. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων για δύο λεπτά, ο κύριος Όμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών για το άσυλο θα έπρεπε να στηρίζεται από τα κράτη-μέλη, ειδικά για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές πιέσεις. Όμως έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι όντως απαραίτητη αυτή η νέα υπηρεσία υποστήριξης. Ίσως καταλήξει να επεμβαίνει υπερβολικά στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. και παρόλο που δείχνει να ενδιαφέρεται για υψηλή προστασία για τους ε, ετούντες άσυλος, ίσως καταλήξει να δημιουργήσει προβλήματα για τις πιο γενναιόδορες χώρες όσον αφορά το άσυλο, όπως στην Αυστρία. Επίσης θεωρώ ότι ο κανονισμός αντιτίθεται στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας που μιλάει για λιγότερες ρυθμίσεις και για επικουρικότητα. Θεωρώ ότι είναι αποσπασματική η προσέγγιση μας για το άσυλο και τη μετανάστευση και ένα από τα αποσπάσματα είναι και αυτός ο κανονισμός. Επίσης, να μεταφέρω και την ακόλουθη κριτική. Μπορεί να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας αν είμαστε υπερβολικά γενναιόδοροι με το άσυλο. Αν επιτρέψουμε και σε άλλες γενιές τι οικογένειε των ετούντων άσυλων να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ άλλων και στην αγορά απασχόληση, τώρα που αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την ανεργία. Και θα εξορδόντω όλο και περισσότεροι από τα επιδόματα ανεργίας πρέπει να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το άσυλο και τη μετανάστευση διαφορετικά δεν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Τελώσαμε τους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων και τώρα έχουν το λόγο οι συνάδελφοι που λαμβάνουν το λόγο ε, για δικό τους σκοπό. Ο κ. Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντική η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και έτσι συμβολικά νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή πραγματοποιείται στη Μάλτα σε μια χώρα του ευρωπαϊκού νότου που δέχεται μεγάλες πιέσεις τόσο από εκείνου που αιτούνται άσυλο όσο και ε, στα πλαίσια των θεμάτων της παράνομης μετανάστευσης. Και είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί, να συντονιστεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και τελικά να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία προσέγγιση ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικές πρακτικές τη στιγμή μάλιστα που όλοι αναγνωρίζουμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. για παράδειγμα και αυτά τα στοιχεία είναι στη διάθεση και της επιτροπής αν νομίζω ότι τα ξέρει ήδη ε, ένας ιρακινός που αιτείται άσυλο ε, σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει πιθανότητες 71% η έτσι αυτή να γίνει δεκτή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος οι πιθανότητες αυτές μπορεί να είναι μόνο 2%. και βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικά προβλήματα ανάμεσα στα κράτη μέλη ε, η συμφωνία δουβλίνο 2 είναι δεδομένο ότι επίσης επιβαρύνει περισσότερο κάποια κράτη μέλη σε σχέση με κάποια άλλα. Ε, και βεβαίως αυτή η υπηρεσία για το άσυλο έρχεται να ε, υποστηρίξει και τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που προσφέρονται και μέσα από το ευρωπαϊκό ταμείο προσφύγων και αναφέρομαι στη μεταφορά και στην επανεγκατάσταση προσφύγων τόσο σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες από τρίτες χώρες στην ευρώπη ε, όσο βεβαίως και στο λεγόμενο reallocation στην ε, εσωτερική επανεγκατάσταση προσφύγων. σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση από τρίτες χώρες κάνουμε βήματα βεβαίω μικρά βήματα αλλά προσπαθούμε. σε ό,τι αφορά όμω και αυτό θέλω να το τονίσω στην αξιότιμη κυρία επίτροπο την εσωτερική επανεγκατάσταση προσφύγων παρά το γεγονό ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα βάρη σε κάποια κράτη μέλη κυρίω στον ευρωπαϊκό νότο σε σχέση με κάποια άλλα δεν έχουμε κάνει καμία ειδική πρόταση δεν έχουμε πάρει καμιά πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά αναμένουμε τις προτάσεις της επιτροπής έχουμε στείλει και σχετική ε, επιστολή ε, στα πλαίσια της επιτροπής libe και αν μη τι άλλο να δείξουμε μεγαλύτερη τόλμη σε αυτά τα θέματα γιατί ε, οι πιέσει είναι πολύ μεγάλε. κλείνοντα κύριε πρόεδρε θέλω να καταλήξω με το εξή είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε του μηχανισμού στην ευρωπαϊκή ένωση για την υποδοχή προσφύγων για την αποδοχή αιτήσεων για άσυλο όχι μόνο για ανθρωπιστικού λόγου και για λόγου που έχουν αναφερθεί ήδη από του άλλου συναδέλφου αλλά και για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. πρέπει να δώσουμε σε όλου εκείνου που ψάχνουν μια καλύτερη πατρίδα ένα καλύτερο μέλλον το μήνυμα ότι στην ευρώπη αναζητώντα κανεί τι νόμιμε οδού έχει καλύτερε πιθανότητε αντί να επιλέξει εκείνε τι παράνομη μετανάστευση που δυστυχώ οι πιέσει είναι πολύ μεγάλε. ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ. Για δυόμιση λεπτά. Για δυόμιση λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριος Μπάφτον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο αντιβαίνει με το opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου προτάσεις για 40 εκατομμύρια προκειμένου ότι για δημιουργηθεί μια υπηρεσία στη Μάλτα έρχεται αντίθετη με τις ε, κρατικές αρμοδιότητες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα που έχουν να κάνουν με τη φύλαξη των συνόρων και τα λοιπά, δεν θα έπρεπε να συζητούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τον πληθυσμό και θα έπρεπε να μπορεί να το ελέγξει. Το Ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις. Αυτά τα 40 εκατομμύρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δημιουργία νέων σχολείων και για να βελτιώσουν ε, την ποιότητα ζωή όλων. Σας υπενθυμίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο μία στις τέσσερις γεννήσεις δεν είναι από μητέρε που έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί δίνονται χρήματα του Βρετανού φορολογούμενου μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Στην ε, προεκλογική εκστρατεία όλα τα πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου λένε ότι θα κάνουν κάτι για την μετανάστευση. Όμως τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς εσάς όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει όλες τις αρμοδιότητες σε θέματα ασύλου. Πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει ότι αδιαφορεί για τις ανάγκες και τις επιθυμίες των Βρετανών πρέπει να έχουμε opt-out και εδώ. Νομίζω ότι οι Βρετανοί χρειάζονται ειλικρίνεια από εσάς γιατί υποτίθεται ότι εσείς τους εκπροσωπείτε και θα έπρεπε να γνωρίζουν τι σχεδιάζετε. Τελειώσαμε με τους εγγεγραμμένους ομιλητές και μπαίνουμε στις ε, παρεμβάσεις ενός λεπτού. Μόνο ο κύριος Σιλβέστρης ζήτησε το λόγο και τον έχει για ένα λεπτό. Θα σας διακόψω όμως πάνω στο λεπτό, να το ξέρετε. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για αλληλεγγύη μόνο έτσι απλά, διότι ένα γραφείο υποστήριξης χρειάζεται μία υποδομή για τους ετούντες άσυλο θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία γρήγορη, ταχεία διαδικασία χορήγησης ασύλου και βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνονται παραβάσεις και παραβιάσεις, καθώς και καταχρήσεις. Θα ήθελα να πω αυτά που είπε και ο κύριος Μποργέζιο. Ε, η Νότιος Ιταλία, Ιταλία δηλαδή, και στη Νότιο Ιταλία ε, το ίδιο αυτό το μέρος θα μπορούσε να θεωρηθεί μία πύλη για την είσοδο μεταναστών. Αυτό αφορά τη Μάλτα, την Νότια Ιταλία και ούτω καθεξής. Αυτές οι περιφέρειες που γυτνιάζουν με τους χώρους υποδοχής θα πρέπει να μας απασχολήσουν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Επίτροπο. και θα κλείσει τη συζήτηση η συγγήτρια Τζιν Jean Lambert. Μάλστρομ, σας ευχαριστώ πολύ γιατί δημιουργήθηκαν, ε, δημιουργήθηκε αυτή η υπηρεσία με μεγάλη πλειοψηφία. Υπήρχε ομοφωνία από όλα τα κράτη-μέλη. Και εμείς δεχόμαστε την ρήτρα αυτοεξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξε όμως μεγάλη υποστήριξη για ένα γραφείο υποστήριξης το οποίο θα δημιουργηθεί. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τρίτες χώρες, ε, εποχικά δηλαδή, και θα μπορέσει να βοηθήσει αυτό το γραφείο, αυτό ο φορέας. Αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχει εισδοχή στο Βορρά, στην ε, Κεντρική Ευρώπη και στο Νότο. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο το ότι βρίσκεται στη Βαλέτα. Δεν πρόκειται για έναν άλλο φορέα. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σύστασης μιας πραγματικής πολιτικής ασύλου, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν πρακτικές και κοινά πρότυπα για τις χώρες που υφίστανται πίεση, να υπάρχει ένας ειδικό τοπος να στέλνονται εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Και μετά τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ποιος θα παραμείνει και ποιος όχι. Χρειάζεται όμως εναρμόνιση των διαδικασιών. Και βεβαίως θα πρέπει να προωθήσουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα τμήμα, διότι όπως είπε και η κυρία Λάμπερτ, το υπόλοιπο πακέτο δεν έχει διευθετηθεί και δυστυχώς δεν υπήρξε υποστήριξη του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα στο εγγύς μέλλον. Για πάση περιπτώσει όχι στο τόσο μακρινό. Το λόγο έχει η Τζιν Λάμπερτ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να δράξω την ευκαιρία για να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν αν και δυστυχώς δεν είναι παρόντες όλοι οι ερωτώντες. Ποιες είναι οι υποχρέσεις για το άσυλο αυτό διευκρινίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις που όλα τα κράτη-μέλη μεμονωμένα έχουν υπογράψει. Αυτό δεν είναι το ίδιο με την πολιτική μετανάστευση και θα έπρεπε να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά. Και για όσους ανησυχούν για τα χρήματα. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις που είναι εθνικές και πολιτικές. Αν κάποια κράτη-μέλη μας σταματήσουν να δημιουργούν πρόσφυγες στο Ιράν και στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα τις κακουχίες πολλών ανθρώπων όσον αφορά κάποια άλλα θέματα. Ελπίζουμε ότι βελτιώνοντας την ποιότητα του συστήματος σε κάποια κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και να ξεμπλοκάρουμε ορισμένα άλλα κομμάτια του συστήματος ασύλου και να βοηθήσουμε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις. Ανέφεραν κάποιοι ότι ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γεωγραφικές πιέσεις εξαιτίας των ροών εισόδου, όμως πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα δεν είναι καν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άκουσα με ενδιαφέρον κάποιον συνάδελφο που ζήτησε περισσότερη υποστήριξη, όμως δεν είδα τις τροπολογίες σας τις σχετικές. Να διευκρινίσω επίσης ότι η Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δεν θα αποφασίζει για την κατάσταση των ετούντων. Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη στο ρόλο αυτό. Οπότε ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ενεργό συμμετοχή τους και για τη βοήθησή τους και ελπίζω ότι όλοι αναμένουμε να παραβρεθούμε στη Βαλέτα όταν θα κοπεί η κορδέλα και θα εγγενιαστεί η υπηρεσία. η συζήτηση. Και δεν πρέπει να, ξεχάσουμε